ΝΑΤΟ για το πολιτές σχέδιο αποκατάσταση του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Ο κύριος Μάτο έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. κύριε Πρόεδρε, αυτή Επίτροπο συζητούμε για την πρόταση που έχει σαν αντικείμενο το σχέδιο αποκα... αποκατάστασης του τόνου στο ε, Ανατολικό Ανθλαντικό και στην ε, Μεσόγειο. Όπως ξέρετε, από το 2016 υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο αποκατάστασης του τόνου, το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2022 και οι Αλείς έκαναν, κατάβαλαν μια τεράστια προσπάθεια για να προσαρμόσουν τα λιεύματά τους στον όγκο το, των μειωμένων αλευμάτων τηρώντας τις αυστηρές αυτές προϋποθέσεις. Και χάρη σε αυτό η βιομάζα του τόνου, η οποία καταχωρήθηκε το 2008, είχε μια ε, θετική ε, τάση και γι' αυτό η ΚΑΤ αποφάσισε να αυξήσει τον όγκο των αλλιευμάτων το 2017 γιατί υπάρχουν δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι τα αποθέματα βρίσκονται σε, ένα, σε μια κατάσταση αυθονίας, υγιούς αυθονίας. Άρα η ανάκαμψη του, των αποθεμάτων του τόνου ε, θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια απόφαση της ΚΑΤ να αυξήσει παραπάνω αυτό τον όγκο και αυτό ακριβώς ζητήσαμε και εμείς. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στους αλληλείς ε, όπως γίνεται στα Κανάρια για παράδειγμα παράδειγμα που ε, ασκούν ε, την βιοτεχνική αλία του, τόνου είναι, του τόνου είναι πολύ δύσκολο να του εξηγήσουμε ότι στις 24 ώρες ε, θα πρέπει να αποσυρθούν εφόσον έχουν καλυφθεί οι ποσοστώσεις. Η νομοθετική πρωτοβουλία την οποία συζητούμε σήμερα ανταποκρίνεται στο στόχο να αγγιηθούμε μια ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτού του προγράμματος αποκατάσταση. Η πρόταση περιλαμβάνει τεχνικά μέτρα όπως ε, ε, τα θέματα του, της αλίευσης του ζωντανού τόνου και την ε, χρήση στεροσκοπικών ε, συσκευών για να εξετάζονται τα αποθέματα και το πρόγραμμα επιθεώρησης που προτείνει η ΚΑΤ. Η Επιτροπή Επιτροπή εφαρμόζει σωστά τις προτάσεις της ΕΚΑΤ και πιστεύουμε ότι πηγαίνουμε ακόμα και πιο πέρα από αυτό το οποίο έχει ήδη αποφασιστεί. Και θα ήθελα να σε ότι ότι ο στόχος ε, εφαρμογής των προτάσεων ΚΑΤ αφορά την ομοιογένεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια νέα συζήτηση για θέματα τα οποία ήδη έχουν αποφασιστεί. Η ε, έκθεση έχει σαν στόχο να εγγυηθεί την ισοτιμία των προϋποθέσεων για όλους όσους συμμετέχουν στην αλία του τόνου και ε, του αλείς των τρίτων χωρών γιατί εάν εφαρμοστούν διαφορετικοί κανόνες για τους αλλοδαπού στόλου, όλες οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και όλοι οι περιορισμοί που έχουν εφαρμοστεί για τους Ευρωπαίου αλείς θα είναι μάτες. Από την άλλη, και αυτό είναι ένα θέμα διαφάνειας, η Επιτροπή προτείνει να εφαρμοστούν οι τροπολογίε μέσω εκτελεστικών πράξεων. Και εδώ ε, δεν είμαστε σύμφωνοι, γιατί πιστεύουμε ότι η εφαρμογή αυτών των συστάσεων θα πρέπει να είναι κοινή αρμοδιότητα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου στο πλαίσιο του, κανον... Ε, τακτού... του συνήθους διαδικασίας και να εμπέπτει στην ε, συναπόφαση. Εγώ πάντοτε ζήτησα το Κοινοβούλιο να έχει την αρμοδιότητα της συναπόφασης και να μην εφαρμόζεται πρακτικές για να συρρυκνούνται η επιρροή του Κοινοβουλίου. Διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι οι συστάσει τη ΕΚΑΤ λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων τρόπων αλεία του τόνου. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε τον ρόλο τη ε, ε, παραδοσιακή αλεία στα Κανάρια, για παράδειγμα, όσον αφορά την διατήρηση των αποθεμάτων. Γι' αυτό θα θέλουμε να δώσουμε έμφαση εδώ όσον αφορά την κατανομή των ποσοστώσεων, ούτως ώστε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ε, παραδοσιακές μορφές αλίας. Ε, κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, συνεισέφεραν με την υποβολή τροπολογιών ούτε ώστε να έχουμε ένα κείμενο το οποίο να είναι ικανοποιητικό για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μάτο. Τώρα θα ακούσουμε τον Επίτροπο Βέλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστήσω τον κύριο Γκαμπριέλ Μάτο. Η Κομισιόν εκτιμά ιδιαίτερα το σχέδιο έκθεσης ε, του κύριου Μάτο. Είναι προφανώς το αποτέλεσμα πολύ καλής αντίληψης των ζητημάτων ε, που αφορούν τον τόνο είναι πολύτιμη συνεισφορά και περιέχει κάποιες σημαντικές προτάσεις για τροποποίηση της αρχικής πρότασης. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε πως η πρόταση αυτή στόχο έχει, όπως ήδη αναφέρθηκε, να μεταφέρει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο μέτρα που έχουν ήδη υιοθετηθεί στην Διεθνή Επιτροπή για την Διατήρηση του Τόνου του Ατλαντικού εγκρίθηκαν το 2014 και ισχύουν για τα κραταμέλη και τις εταιρείε από τον Ιούλιο του 2015. Πρέπει να πούμε πως το σχέδιο αυτό αποκατάστασης ε, έχει αναγνωριστεί ως επιτυχία και τα αποθέματα των βρίσκονται σε πορεία αποκατάστασης του των λεχθέντων δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης. Πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στην βιώσιμη διαχείριση του σημαντικού αυτού πόρου. Τα μέτρα που έχουν εγκριθεί στο σχέδιο αυτό από την ICAT λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πολλές από τις διατάξεις του σχεδίου αυτού αποκατάστασης ε, έχουν άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη. Όμως ε, χρειάζεται να υπάρξει μεταφορά στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο για να είναι εφαρμόσιμα αυτά τα μέτρα σε νομικά και φυσικά πρόσωπα και για να υπάρχει συμμόρφωση της Ένωσης με τις διεθνείς υποχρεώσεις της και βεβαίως για να διατηρηθεί η αξιοπιστία της Ένωσης όσον αφορά την αηφόρο διαχείριση αλλιευμάτων. Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση αυτή ανταποκρίνεται σε γενικές γραμμές στις προσδοκίες μας, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποιες αποκλήσεις. Αυτό ισχύει ε, όσον αφορά την ερμηνεία των αρμοδιοτήτων των ε, θεσμικών οργάνων ε, όσον αφορά την μεταφορά διατάξεων από τους τοπικούς οργανισμούς διαχείρισης. Όμως θεωρούμε πως μπορούν να λυθούν όσον αφορά τις διατάξεις τώρα για τον αποκτήσει η Κομισιόν την ικανότητα να εκδίδει πράξεις κάθε εξιοδότηση. Η Κομισιόν θεωρεί πως λόγω των ε, τροποποιήσεων ε, του σχεδίου στην ΑΕΚΑΤ αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της πρότασης. Γιατί, γιατί οι πράξεις κατά εξιοδότηση απαιτούνται για να μπορούμε να δράσουμε γρήγορα και να ενσωματώσουμε μελλοντικέ αλλαγές του σχεδίου αποκατάστασης που θα γίνουν στο επίπεδο της Επιτροπής ΑΕΚΑΤ. Οι τροποποιήσεις αυτές ε, λαμβάνουν χώρα τακτικά και είναι βέβαιο ότι θα συμβούν και αν ακολουθήσουμε την τακτική νομοθετική διαδικασία δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα εγκαίρως για να συμμορφωθεί η Ένωση με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Η έγκριση των πράξεων αυτών κατεξιοδότηση μας δίνει την δυνατότητα να μεταφέρουμε επακριβώς και γρήγορα τις διατάξεις αυτές με το να τροποποιούμε μόνο τα δευτερεύοντα στοιχεία των νομοθετικών πράξεων κατά το οποίο απαιτεί βεβαίως και την κατάλληλη διαβούλευση και διαβούλευση σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Επίσης απαιτεί έγκαιρη μετάδοση των εγγράφων αυτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Κομισιόν επίσης θεωρεί πως θα πρέπει να αποκτήσει την δυνατότητα να εγκρίνει εφαρμοστικές πράξεις, καθώς υπάρχει συχνά η ανάγκη να δούμε πώς θα πρέπει να εφαρμόζονται κάποια μέτρα του σχεδίου αυτού αποκατάστασης στο επίπεδο της Ένωσης. Αυτό χρειάζεται για να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα μέτρα ελέγχου που εισάγονται στην ΆΕΚΑΤ όπου η ερμηνεία μπορεί να διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και σχετίζονται άμεσα με το σεβασμό των ποσοστώσεων και άλλων διεθνών υποχρεώσεων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, η πρόταση της Κομισιόν για έναν κανονισμό για το πολιετές σχέδιο αποκατάστασης ε, του τόνου μας, ε, μας δίνει την ε, ε, δυνατότητα εφαρμογής αυτής της συμφωνίας και όπως είπα πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή συνεισφορά η έκθεση του κυρίου Μάτου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Επίτροπε και τώρα ξεκινάμε τη συζήτηση με τις πολιτικές ομάδες. Πρώτος ο κύριος Βαλέσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μάτο και να στηρίξω αυτή τη νέα πρόταση που στόχο έχει την ε, μεταγραφή των ευρωπαϊκών μέτρων για, όπως υιοθετήθηκαν από την ΙΚΑΤ για την ε, ανάκαμψη των στόκ ε, του τόνου στον, Ατλαντικό, στον Ανατολικό Ατλαντικό. Θα πρέπει να γίνουν δύο βήματα. Καταρχήν θα πρέπει να αυξηθούν τα συνολικά επιτρεπόμενα λιεύματα, τα ΤΑΚ, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ε, προσεκτική όσον αφορά την αλίευση σε συγκεκριμένες περιοχές, τους χρόνου, τη περιόδου αλίευση αλλά και τα μήνυμα μεγέθη. Να ενισχύσουμε το σχέδιο της ΕΚΑΤ για ε, κοινού διεθνεί ελέγχου. Θα πρέπει όντω ε, ο κανόνας αυτός να ισχύει ομοιόμορφα για να εξασφαλιστεί ισότιμο ανταγωνισμό και συμπεριλαμβανομένων των μη ευρωπαϊκών ε, φορέων και αλλιών. Εάν συσχίσουν διαφορετικοί κανόνε για του ξένου τους ξένους τους ενώ ισχύουν όλοι αυτοί οι περιορισμοί, δεν θα έχουν καν αποτελέσματα οι περιορισμοί για του Ευρωπαίου αλλιεί και θα φανεί ότι εμεί τιμωρούμε του δικού μα αλλιεί. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα του επιβάλλουμε αυστηρότερα μέτρα Γι' αυτό θέλω... Και τέλος θα στηρίξω την ε, εργασία του κυρίου Μάτο για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Μπριάνο, 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε. Σήμερα δεν θέλω μόνο να μιλήσω για την αποδοχή των συστάσεων ΙΚΑΤ επί των οποίων συμφωνούμε και μάλιστα με τον κύριο Μάτο που είναι εισηγητή, το έχουμε ευρύτατα συζητήσει το θέμα ανάμεσα στι ομάδε, στην Επιτροπή Αλληγία. αλλά κατά τη γνώμη μου έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τον τόνο τόσο όσον αφορά την οικολογία του είδου, δηλαδή αποκατάσταση των στόκων όσο και κοινωνικο οικονομικού τομεί, που που συνδέονται με την αλληλεία του τόνου. Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κράτη-μέλη είναι συμβαλόμενο μέρος της ΣΥΚΑΤ. Και το 2014 ε, στην Γένοβα, που είναι και η πόλη μου μάλιστα, στην ετήσια σύνοδο της ΣΥΚΑΤ, θετικά δεχτήκαμε το νέο για τα θετικά στοιχεία, για την καλή υγεία των στόκων του τόνου και τότε να αποφασίστηκε και το 21% αύξηση των ποσοστώσεων που αποδίδονται στις συμφιλόμενα κράτη. Οι ποσοστώσεις ορίζονται από την ΙΚΑ, αλλά τα κριτήρια κατανομής αποφασίζονται από τα κρατημέλη. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις αυτές τις ποσοστώσεις ωφελούν μόνο λίγοι ε, εφοπλιστές, ενώ οι βιοτέχνες αλληλεί διαρκώς αποκλείονται παρά την αύξηση αυτού του 20%. Χωρίς να ξεχνάμε ότι αν τυχαία αλλιευθεί ένας, ένα τόνος, ο μικρός αλλιές μπορεί να τιμωρηθεί πολύ αυστηρά. Θα ε, περίμενα λοιπόν μια πιο ισότιμη κατανομή Γι' αυτό και οι σοσιαλιστές έχουν υποβάλει μια τροπολογία που, κατα... καταγγέλει τον μηχανισμό του μονοπωλίου των μεγάλων εφοπλιστών και που ζητά από τα κρατήμερα να... να θεωρήσουν πιο ισότιμα την κατανομή των ποσοστώσεων αλληλείας του τόνου. Ευχαριστώ. Τόμα, έτσι ένα λεπτό. Σήμερα η αλληλεία ως οικονομική δραστηριότητα εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ κοινωνικής βιωσιμότητας των ε, στόλων και διατήρηση των αποθεμάτων. Ιδιαίτερα οι θαλάσσιοι πόροι έχουν ε, καθαριστική σημασία ε, ωστόσο από την άλλη και η αλείς θα πρέπει να διαφυλάξει το δικό της οικονομικό συμφέρον ε, παρά τους περιορισμούς στην Αλία και θεωρώ ότι η έκθεση αυτή αναγνωρίζει την ανάγκη αυτής της ισορροπίας και πραγματικά είναι τιμή μου που είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στην έκθεση αυτή ε, Στη συνέχεια με τον κύριο Μάτο και τους Σκιώδης μετά την ε, ανασύσταση ε, των αποθεμάτων του ερυθρού τόνου ε, τελικά έχουμε την ευκαιρία να αυξήσουμε τις ποσοστώσεις για το 2016 αυξάνοντας και τα κέρδη για τους αλλοίς που αλλιεύουν παραδοσιακές μεθόδους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μάτο. Και θα ήθελα να πω ότι στηρίζουμε αυτή την έκθεση γιατί εμβαθύνει στο σχέδιο ανασύσταση των αποθεμάτων ερθρού τόνου στη Μεσόγειο στη βάση επιστημονικών ε, δεδομένων. Η εξέλιξη της ε, βιομάζας το επαληθεύει. Ε, το 2012 ε, είχαμε μια απώλεια της ε, αλληλευτικής ε, ικανότητας πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο οι στόλοι οι οποίοι αλλιεύουν στην ε, Μεσόγειο, είτε οι ευρωπαϊκοί είτε οι στόλοι των τρίτων χωρών, να εργάζονται υπό ισότιμες προϋποθέσεις. Δεν είναι δυνατόν ε, να ζημιώνονται οι αλλοί των τρίτων χωρών όταν ε, αποτεχάνουν οι συμφωνίες. Και τελικά ισχύει για όλους η προσπάθεια διαφύλαξης του οικοσυστήματος. Ε, εμείς ε, στα Κανάρια νησιά είμαστε υπέρ ε, της διαφύλαξης παραδοσιακών τεχνικών παγίδευσης του τόνου. Αλλά δεν συμφωνούμε με, εξ, εκφράσεις που ποινικοποιούν ε, τους αλείς επειδή εφαρμόζονται κάποιε αθέμητε αληφτικέ ε, πρακτικέ. Υποστηρίζουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου όσον αφορά την μεταφορά των συστάσεων των ε, περιφερειακών οργανώσεων αλλίε, γιατί πραγματικά ε, εισφέρουν στην αύξηση τη διαφάνεια το θέμα της, ε, τα προβλήματα της αλίας ε, είναι μια ένταξη ότι συμβαίνει όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση απομακρύνεται από τον πολίτη. Ε, γι' αυτό σας παρακαλούμε να, στηρίξετε στη, να στηριχθείτε στη δική μας συμμετοχή. Κυρία Χαζακάμπ, ευχαριστώ. Ο ερυθρός τόνος είναι ίσως το πιο γνωστό αλίευμα που γνωρίζουμε. Κάτι βεβαίως το οποίο δεν το βοηθάει ιδιαίτερα. Έχει πέσει σε ένα διάστημα 50 ετών το απόθεμα του αλεύματος κατά 90 σχεδόν της 100. Ε, στην αρχή βεβαίως είχαμε επί δεκαετίες ε, τρομερή υπεραλίευση η οποία όφιλόταν ε, στην επιδοτούμενη υπερβολική δυναμικότητα του Ευρωπαϊκού Στόλου. Το 2006 ελήφθησαν κάποια μέτρα για να περιοριστεί η υπεραλία και να προστατευτεί ο τόνος, αλλά Βεβαίω, όσο και αν από ό,τι φαίνεται λειτουργούν τα μέτρα, δεν έχει φτάσει ακόμα η στιγμή για να χαιρόμαστε. Ο τόνος είχε φτάσει σχεδόν στο μηδέν και μετά διπλασιάζεται ε, το απόθεμα. Ε, Παρ' όλα αυτά έχουμε κινήσει από πάρα πολύ χαμηλή βάση και πάρα πολλές ε, οργανώσεις προειδοποιούν ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να ξαναρχίσουμε να ψαρεύουμε περισσότερο τόνο. Και αυτό ακριβώς θέλει ο εισηγητής και η Κομισιόν, περισσότερη αλληλεία. Και δεν ε, συμφωνούμε βεβαίω και για το παραλίευμα ε, άλλων ειδών, τα οποία μετά τα πετάμε γιατί ο στόχος μας είναι ο τόνος. Κυρία Πρόεδρε, το κόμμα των ζώων δεν θα υπερψηφίσει αυτή την έκθεση γιατί θεωρούμε πως ε, έτσι διαγουμίζουμε τον πλανήτη και θεωρούμε πως θα πρέπει να τελειώσουν οι επιδοτήσεις προς την Αλία και τη Γεωργία. Thank you. Mr. one minute. ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αντιπροσωπεία μας είναι υπέρ της έκθεσης αυτής, επί της οποίας εργαστήκαμε μαζί με τους συναδέλφους και με τον ε, κύριο Μάτο, γιατί είναι σημαντικό να λαμβάνουμε τις υποδείξεις της ΣΥΚΕΤ που έχουν λειτουργήσει εξάλλου σωστά τα τελευταία χρόνια και είναι σημαντικό αυτό να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μέχρι τον περασμένο αιώνα, μόνο με τον παραδοσιακό τρόπο αλλιώ ο τόνος, μετά έγινε βιομηχανία και μετά κατέρευσε ε, ο αληφτικός πόρος. Φαίνεται πως η αποκατάσταση σε λειτουργεί και η Επίτροπε Βέλα και άρα είναι σωστή η πορεία αυτή. Αν και, ανησυχη... Αν και συμμερίζομαι την ανησυχία ορισμένων που λένε ότι είναι πρόημο το να αυξηθούν οι ποσοστώσει. Λειτουργούν οι ποσοστώσει για το περιβαλλοντικό τομέα, αλλά όχι για το κοινωνικο-οικονομικό. Η κοινωνική δικαιοσύνη έχει μείνει περιφερειακή, μάλλον περιθωριακή υπόθεση, η βιοτεχνική δηλαδή ε, αλληλεία. Ακόμα και αν δεν μα αρέσει πολύ η φόρμα που παρουσίασε την τροπολογία η κυρία Βιάνο, θα την υποστηρίξουμε γιατί πιστεύω πω θα πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Ε, ίσως είναι ένα πρόβλημα που ίσως να μην είναι ο κατάλληλος χώρος για να το συζητήσουμε, όμως το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να ε, εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να κάνει τη φωνή του ακουστή και για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κυρία Ροντούστο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, μεγάλα ψάρια με μικρή κλίμακα σαλίας Αυτό είναι εφικτό για τον τόνο στον ε, Ανατολικό, ε, στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Η βιοτεχνική αλία έχει καλή φήμη όσον αφορά την επιλεκτικότητα καθώς και τις επιπτώσεις για την, στο θαλάσσιο οικοσύστημα που είναι θετικές και την μειωμένη χρήση ενέργειας. Εμείς ε, θεωρούμε ότι η παραδοσιακή αλής θα πρέπει να έχουν επαρκής ε, ποσοστώσεις. Βάσει του κανονισμού η κάθε χώρα μέλος ε, αποφασίζει για τις δικές της αλληλευτικές δυνατότητες πώς κατανέμει στο δικό της αλληλευτικό στόλο. Εδώ θα πρέπει να εφαρμόζονται ε, διαφανή κριτήρια, αλλά όχι μόνο αυτό. Οι τεχνικές αλλήλευσεις με υψηλής επιλεκτικότητας και χαμηλής ενέργειας θα πρέπει να προκρίνονται. Ε, θα πρέπει ε, η όθηση η οποία δίδεται εδώ να συνεχίσει ούτως ώστε να ε, υπάρξει σωστή συμμετοχή της αλίας μικρής κλίμακας της ποσοστώσης. Γιατί πολύ συχνά διαπιστώνονται κρούσματα λοιπούς διαφάνειας στο σύστημα κατανομής των ποσοστώσεων. Γι' αυτό χαιρετίζω την ε, υποχρέωση ε, δήλωσης ε, στοιχείων εκ μέρους των χωρών μετλών. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χοκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύρια Πρόεδρε, ο ερυθρός τόνος είναι ένα δώρο της φύσης και κάποιοι το αποκαλούν ε, ένα χρυσορυχείο που κολυμπάει. Πρέπει λοιπόν να ε, επιζήσει αυτό το είδος και τελικά τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα γιατί το είδος αυτό εξακολουθεί να κινδυνεύει. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποχρέωση να σκεφτεί το πώς θα εφαρμόσει τους ε, κανονισμούς για το πολυετές σχέδιο αποκατάστασης ε, του ερυθρού τόνου. Κάποια πράγματα τώρα εδώ πέρα. Ε, νομικές υποχρεώσεις και τέτοιοι κανονισμοί πρέπει να είναι ξεκάθαροι και να μην επιδέχονται ερμηνείας. Και βεβαίως ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί το εξής αυστηρά για όλους και για τους εκτός της Ένωσης Τρίτων καταπολέμηση της ε, λαθραλίας έχει μεγάλη σημασία. Σας ευχαριστώ. Λόπες Μπερμέχο για λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ε η έκθεση αυτή ε, κάνει ρητή μνήμα στην παραδοσιακή τεχνική της παγίδευσης του τόνου και πραγματικά είναι σημαντικό βήμα στην αναγνώριση αυτής της αλληλευτικής μεθόδου για μια βιώσιμη, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης αλίας. Ε, γιατί είναι σημαντικό για την ε, διατήρηση επίσης των ε, κοινοτήτων των αλλιέων καθώς και για τη διατήρηση του οικοσύστηματος αυτή η έκθεση απευθύνει μια προειδοποίηση σε κυβερνήσει όπω είναι η Ισπανική, κυβέρνηση, η Ισπανική κυβέρνηση, η οποία έχει περιθωριοποιήσει μέχρι στιγμή τι παραδοσιακέ τεχνικέ παγίδευση του τόνου, καθώ και την ε, εθνική κατανομή ε, ποσοστώσεων. Ε, ελπίζουμε η έκθεση αυτή να χρησιμεύσει ούτως ώστε να προθεθεί αυτή η αλληλευτική μέθοδος η οποία είναι βιώσιμη ως προς τις κοινότητες των αλλαίων όσο και ως προς τη διατήρηση του οικοσυστήματος των θαλασσών μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φάρα. Ευχαριστώ. Απόψε μιλάμε για το καταστροφικό επίπεδο στο οποίο έχουν φτάσει τα αποθέματα των Κανείς όμως δεν έχει αναφέρει το ψάρεμα με πετονιά. Έχουμε ένα σύστημα ποσοστώσεων κάτι το οποίο σημαίνει επί δεκαετίες απορρίψεις των άλλων ειδών, των παραλιευμάτων. Θέλουμε λοιπόν έναν εμπορικό τομέα, αλλά δεν υπολογίζουμε το πώς η αλληλεία αναψυχής με πετονιά μπορεί να βοηθήσει αυτόν τον κλάδο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι ψαράδες ε, που ψαρεύουν με πετονιά πέστροφες ε, αποδίδουν στην οικονομία πολύ περισσότερο από, τις, ε, από την εμπορική αλληλεία και στις ε, είπα το ίδιο είδος ε, πλέον θεωρήθηκε από εμπορικό είδος το οποίο μπορεί να λιεύεται σε αλληλεία αναψυχής και πλέον όλες ε, οι αυτές οι κοινότητες στην ανατολική ακτή του Ατλαντικού με την πέστροφα αυτή κατάφεραν να ζουν από τα λευτικά σκάφη κτλ. Και εμείς ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε το γελίο όριο του ενός ψαριού ανά ψαρά και οι αλληλείς βεβαίως ε, οι επαγγελματίες ε, έχουν ένα τελείως δυσανάλογο όριο. Αυτό το κάναμε εσείς το κάνατε ένας Μαλτέζος γραφειοκράτης χωρίς να συζητηθεί από τους υπουργούς ούτε από το κοινοβούλιο και οπωσδήποτε δεν συζητήθηκε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και οι απλοί ερασιτέχνες ψαράδες θα γίνουν εγκληματίες αν κάνουν αυτά τα οποία πάντα έκαναν. Μιλάμε για 800.000 ερασιτέχνες ψαράδες που λένε στο καλό να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς θα φροντίσουμε να συμβεί αυτό. Um, Κύριε Φάρατζ, υπάρχει μια μπλε κάρτα από τον κύριο Κόρμπι. Τη δέχεστε? Παρακαλώ λοιπόν. Κύριε Φαράζ, όπως ξέρετε η κοινή ελληνική πολιτική μεταρρυθμίστηκε πρόσφατα, κάτω το οποίο ακόμα και η Greenpeace ε, χαιρέτησε. Ε, τότε εσείς ήσασταν μέλος και σε δυόμιση χρόνια είχατε πάει σε μία ή δύο συνεδριάσεις όταν ε, συζητούνταν αυτά τα ζητήματα και δίνονταν μεγάλες μάχες. Δεν θεωρείτε λοιπόν πως ε, θα ήσασταν κάπως πιο αξιόπιστος αν είχατε πατήσει ποτέ και στην Επιτροπή Αλληλείας. Well, nice but... Καλή προσπάθεια κύριε Κόρμπατ. Δεν ακούγατε όμως. Ε. Εγώ Εάν πήγαινα σε κάτι στην Επιτροπή Αλία όλα τα χρόνια που ήμουν στο Κοινοβούλιο, δεν είμαι μέλο πλέον, αλλά ακόμα και αν πήγαινα, τίποτα δεν θα μπορούσα να είχα κάνει, ούτε ώστε να βοηθήσω περίπου 800.000 ανθρώπου από τη χώρα μα, οι οποίοι πηγαίνουν να ψαρέψουν. Παρέχουν θέσει εργασία στι παράκτιε κοινωνίε. Δίνουν δουλειέ όσον αφορά εκεί που φτιάχνουν δολώματα, καλάμια κλπ. Πραγματικά δίνουν σημαντικό υπόβαθρο για τα λιμάνια και τι παράκτη κοινότητε. Και αυτή η απαγόρευση, αυτή η απαγόρευση ήρθε χωρί καν να συζητηθεί στην Επιτροπή Αλίας. Λοιπόν, τι νόημα είχε να πάω στην Επιτροπή Αλίας χωρίς να συζητηθεί το θέμα και να ψηφιστεί στο Κοινοβούλιο. Το έκανε ένας κανονισμός αυτό, το οποίο τον πρόθεσε ένας Μαλτέζος γραφειοκράτης που δεν μπορούμε να ψηφίσουμε γι' αυτόν όταν θα βγάλουμε τη θέση του. Αυτό που θέλει και ο Κόρμπετ είναι να έχουμε σωστή λειτουργούσα δημοκρατία και τότε μπορούμε να συζητούμε πώς θα καταφέρουμε να χειριστούμε τα αποθέματα της Βρετανίας. Λοιπόν, καλή προσπάθεια φίλε μου, αλλά ατύχησες. Αυτό εδώ σταματάμε, ζητώ συγγνώμη σηκώσατε τη γαλάζια κάρτα σας, πήρατε την απάντησή σας, θα σταματήσουμε εδώ και να πάμε στον επόμενο αγωρίτη. Την κυρία Αγιέρα Γκαρσία που έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνούμε με την έκθεση αυτή του κυρίου Μάτο για την εφαρμογή της ε, σύστασης για την αλία. Όλα τα σχέδια όμως με κάποια εξαίρεση θέλω να υπενθυμίσω τόνισαν δύο θέματα ουσιώδη και θέλω και εγώ να ενταχθώ σε αυτή τη συζήτηση με την παρέμβασή μου. Ένα θέμα, ενιαία εφαρμογή και αποτελεσματική εφαρμογή από όλους όμως. Και αυτό που συμβαίνει και πικρίνουν οι αλληλείς είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτή την ε, εφαρμογή την ε, ακολουθούν, όχι όμως τα τρίτα, ε, οι τρίτες χώρες και αυτό δημιουργεί προβλήματα στη Μεσόγειο. Σημειώστε λοιπόν επίσης Επίτροπε έχουμε και το θέμα της ανάκαμψης ε, του τόνου και χαίρομαι γι' αυτό. Όμως ε, της βιοτεχνικής αλληλείας οι αλληλείς ε, υφίστανται προβλήματα και δεν ανακάμπτουν. Πρέπει να σταματήσει το μονοπόλιο σε σχέση με τον ερυθρόπτερο τόνο στα κράτη-μέλη. Και πρέπει να δούμε στην Ισπανία δεν επωφελούνται οι μικροί αλληλείς με τις βιοτεχνικές μορφές αλληλείας όπως την Αλμαντράβα για παράδειγμα. Κύριε Βαντάλεν, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα συζητάμε το θέμα αυτό των μέτρων, των μέτρων για την αλληλεία του τόνου. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της όλης διαδικασίας που ακολουθείτε. Νομίζω ότι από πλευρά εισηγητού υπήρξε σωστή αντιμετώπιση, σαφής, θα γίνουν κάποιοι τριμερείς διάλογοι και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού. Ελπίζω να είναι θετική εξέλιξη. Αυτό από τη μια. Από την άλλη πλευρά ανησυχώ τα μάλα για άλλα είδη ψαριών στη Μεσόγειο. Τι θα γίνει με αυτά. Σχεδόν όλα τα είδη υπεραλλιεύονται στην ε, Μεσόγειο. Παίρνω σχάρι ένα είδο γάδου που ε, ψαρεύεται 10 φορές παραπάνω ε, και Επίσης και, τους, ε, και τα νέα ψάρια αλλιεύονται και το ίδιο ισχύει και, για τα, και το γόνο των ψαριών αλλιεύουν και το ίδιο ισχύει και για άλλα είδη. Λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συντάξει ένα σύστημα συντήρησης για το γάδο στην ε, Μεσόγειο αλλά όταν ε, θεσπίζεται φόρο για τη Μεσόγειο εστέ πιο φιλόδοξη για να καλύψετε επίσης όλα τα είδη, όχι μόνο ένα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σεράος Σάντου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Είναι πάντα χαρά να σας έχουμε ανάμεσά μας. Ε, θέλω να χαιρετήσω επίσης τον εισηγητή Γκαμπριέλ το Έκανε σημαντική δουλειά και αναφέρει στο Κοινοβούλιο ένα σύνολο αποφάσεων που όπως αναφέρεται έχουν μεγάλη σημασία στη συζήτησή τους. Για την ενίσχυση της τροποποίησης αυτής ε, από τους σοσιαλδημοκράτες τονίζουμε την ε, προοπτική να καταπολεμηθούν τα μονοπόλια στην Αλία. Παρόλη την εσωτερική κατανομή ποσοστώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θα πρέπει θετικά να επωφελήσουν την βιοτεχνική αλία όπως στις ε, υπερπεριφερειακές περιοχές ασκείται και να μην ε, ε, οδηγήσουμε σε ασφυξία αυτή την αλία στις υπερπεριφερειακές περιοχές όπως στις Αζόρες. Επαναλαμβάνω την ανάγκη να συσσεβαστούμε τις επιστημονικές συστάσεις και να χρησιμοποιήσουμε με σύνεση την αρχή της πρόληψης. Στην αλληλεία του τόνου συνεχίζουν να υπάρχουν υπερβολικές υπερβολικές διατάξεις όσον αφορά την συμπίκνωση της προσπάθειας αλίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αρχίζουμε τη δικασία του Catch the Eye, προσέλκυση προσεχής του Προέδρου. Ο κ. Καπούτο είναι ο πρώτος που έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα σταθώ σε δύο σημεία και μόνο. Το πρώτο αφορά το θέμα των κατηγοριών πράξεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τι μεθοδικέ τροποποίησει του σχεδίου τη αποκαταστάσεω του ρηθρού τόνου στον Ατλαντικό, τον Ανατολικό και στη Μεσόγειο μέσω άρθρων κατοξιδότηση. Αυτόν συμβεί στην πραγματικότητα το Κοινοβούλιο δεν θα έχει πλέον κανένα λόγο και δεν μπορεί να επηρεάσει την όλη κατάσταση. Κατά την άποψή μου, η αποδοχή τη συστάσεω των διαφόρων οργανώσεων των περιφερειακών τη διαχείριση αλληλεία θα πρέπει να παραμείνει μια αρμοδιότητα κοινή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στα πλαίσια τη διαδικασία τη τακτική συναπόφαση. Το δεύτερο σημείο αφορά τι ποσοστώσει για την αλληλεία του ρηθού τόνου. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει ποικιλία ποσόστοση για κάθε σκάφο και αφορά μόνο την, το αλίευμα του 2000 και πώ τέτοια ποσόστοση εκ των πραγμάτων μπορεί να είναι υποφελή για κάποιου αλληλεί και επιζήμια πολλού άλλου φορεί, κυρίω μικρού αλληλεί. Θα πρέπει λοιπόν να απελευθερώσουμε το μηχανισμό των ποσοστώσεων αλληλεία θεωρηθού τόνο από το μονοπόλιο των μεγάλων εφοπλιστών, ευνοώντα πιο βιώσιμη αλληλεία υπέρ των μικρομεσών επιχειρήσεων. Σαν ομάδα SND είχαμε προτείνει κάποια τροπολογία για να καλέσουμε τα κρατημέλη και να επανεξετάσουν το παρόν σύστημα και στους συναδέλφους να υποστηρίξουν το κίνημά αυτό, την κίνησή μα αυτή μας. Ο κύριος Μαρία έχει το λόγο. Η αλία του τόνου στη Μεσόγειο αλλά και στον Ατλαντικό είναι ιδιαίτερη σημασία καθώ πέραν των άλλων συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασία σε πολλέ χώρε εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2006 η ΆΕΚΑΤ θέσπισε ένα πολιετές πλαίσιο που λύγει το 2022 με στόχο την αποκατάσταση του τόνου ώστε να ανασυσταθούν τα αποθέματα τόνου στον ατλαντικό και τη μεσόγειο. κύριε επίτροπε κύριε Βέλλα, στην ελλάδα οι αλληλείς έχουν υποστεί τεράστια ζημιά από το μνημόνιο. μάλιστα από σήμερα κλιμακώνουν τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις ενάντια στη φορομπηχτική λαιλασία και στο αντιασφαλιστικό ρεσάλτο στα πενιχρά εισοδήματά τους αποκλείοντας το λιμάνι του βόλου και τη νέα μηχανιώνα στη θεσσαλονίκη στο πλευρό τους και οι αλλοί του παγκαίου της κρήτης της φθιώτιδας ετοιμάζουν θερμό γενάρη ενάντια στην τρόικα και τους δανειστές. οι έλληνες αλλοί δεν πρόκειται να δεχτούν το αγροτικό μνημόνιο που διαλύει τη ζωή τους τις οικογένειές τους τις επιχειρήσεις τους. απαιτούν δίκαιη ανταμοιβή του κόπου τους απαιτούν ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα και θα παλέψουν ενωμένοι με βάση τα δίκαια αιτήματά τους για την ίδια τους την επιβίωση. ευχαριστώ. Uh, Νομίζω ότι υπήρξε ένα πρόβλημα με, την, με το σύστημα της διαρμηνίας, αν μπορεί να επιλύσει. Κυρία Τζουφρίδα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαστε ικανοποιημένοι διότι χάρη στην προσοχή και στα διάφορα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΙΚΑΤ το πολύτιμο είδος του ερυθρού τόνου εκ νέου ε, αυξάνεται στις θάλασσές μας. Ένα είδος είναι πάρα πολύ πολύτιμο σε όλες τις έννοιες διότι και εμπορικά αποτελεί σίγουρα στην Μεσόγειο ε, αντικείμενο μονοπωλίου δυστυχώς όμως. Έχουμε την περίπτωση αυτό που συμβαίνει στη Σικελία. Μεγάλοι εφοπλιστέ εκμεταλλεύονται την ροή τη μεταναστευτική, ούτω ώστε να βάλουν στα δίκτυα του του τόνου που μπορούν μετά να διατεθούν στο εμπόριο στην Ιαπωνία. Τα αποτελέσματα είναι ότι τώρα ο τόνο, ο οποίο καταφθάνει στα τραπέζια μα, προφέρεται από τον ελληνικό. Είναι με, το κίτρινο πτερίγιο. Ενώ οι Σικελοί αναγκάζονται να εκφορτώσουν τα σκάφη του. Θα πρέπει να προστατεύσουμε του μικρού αλληλεί και τι παραδοσιακέ τεχνικέ. Τα παλιά συστήματα που είναι βιώσιμα που σιγά σιγά όμω εξαφανίζονται. Είναι μια κληρονομιά που θα πρέπει να προστατευτεί διότι είναι πολύτιμη η αλληλεία του ρυθμού τόνου με τον παραδοσιακό τρόπο. Ευχαριστώ. Κύριε Γιάκοφτσεκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο γαλάζιος τόνος ε, είναι ένα είδος ε, προς εξαφάνιση και παρόλο που υπάρχουν κάποια θετικά παραδείγματα όσον αφορά την ανάκαμψη του είδους αυτού των αποθεμάτων και είχαμε κάποια θετικά στοιχεία που είδαμε προσφάτως και προσπαθούμε να αυξήσουμε τις ποσοστώσεις παρόλα αυτά θα ήθελα να καλέσω την ποιή και εσάς κύριε Επίτροπε να είσαστε προσεκτικοί. Ο γαλάζιος τόνος ε, είναι ένα είδος ε, που τελεί υποκίνδυνο και ο τρόπος ε, με τον οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα αλλιεύματα, αυτά τα αποθέματα πρέπει να αναλυθεί, κυρίως όσον αφορά τον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο. Δεν θέλουμε τα μεγάλα μονοπόλια να επικρατήσουν και να κάνουν τη δουλειά τους όπως πάντα. Πιστεύω ότι αυτό θα μας φέρει την ίδια κατάσταση εκ νέου, όπως παλιά. Άρα, χρειαζόμαστε μια αναθεώρηση της καταστάσεως, μια αποτίμηση όλων των αποθεμάτων και στον Ατλαντικό και στην Μεσόγειο. Κύριε Φερέιρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Το πολιτές ε, πρόγραμμα για την ανάκαμψη των ελληνικών είχε θετικές επιπτώσεις σε σχέση με αυτές τις λειτουργικές ενότητες. Ε. Σε σχέση με τη θετική αυτή τάση από το 2008, το 2014 η Διεθνής Επιτροπή για την Αποκατάσταση του Τόνου στον Ατλαντικό οδηγήθηκε στο να πει ότι υπήρξε η αύξηση κατά 20% στα 2015-2016. Από πλευρά μα, ε, με κριτικό πνεύμα ε, αντιμετωπίζουμε τις επικρίσεις ε, όσον αφορά τον τομέα που πλήττει τη βιοτεχνική αλληλεία υπέρ των μεγάλων εταιριών αλληλείας. Και ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιοτεχνική αλληλεία που χρησιμοποιείται στο νότο τη Πορτογαλίας και στην Αλγκάρβη είναι σημαντικό να διασφαλιστεί. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι οι νησιωτικοί αλλήλει που χρησιμοποιούν τέτοιου είδου βιοτεχνική αλληλεία δεν μπορούν να αλλιεύουν σήμερα. Παρότι έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα τη βιοτεχνική αλληλείας. Ιδιαίτερα συλλαμβάνονται τα αλλιεύματα αυτά από άλλου. Στι Αζόρε μόνο μερική αντιστάθμιση, υπάρχει όσον αφορά την αυθύση, την μείωση αυτών των αλλιευμάτων. Ευχαριστώ. Ο κ. Σόλτος είναι ο τελευταίος ομιλητής. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τα μέτρα τα οποία συζητούμε αποτελούν μια συνέχεια. Συνέχεια προσπάθειας διατήρησης των αποθεμάτων του γαλαζοπτέρυγου ε, τόνου. Θα πρέπει να υποθεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε μια εναρμονισμένη προσέγγιση. Εναρμονισμένη όσον αφορά τους διεθνείς κανονισμούς και καθώς αναφορά και τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πρέπει να προστατεύσουμε και τους Ευρωπαίους αλείς. Πρέπει να δοθεί προσοχή σε κάτι που βλέπουν να συμβαίνει συχνά και κάτι που έχει συμβεί για κάποια είδη. Έχουμε τεράστια μονοπόλια. Μονοπόλια τα οποία ε, κινούνται στην αγορά και εκτοπίζουν τους αλληλείς, τους παραδοσιακούς που χρησιμοποιούν παραδοσιακέ μεθόδου, που είναι και οι πιο βιώσιμε. Κάθε κράτο μέλο πιστεύω ότι έχει δυνατότητα να μοιράσει τι ποσοστώσεις στους αλληλεί. Το σημαντικό εδώ είναι ο έλεγχο και η υποβολή αναφορών και ούτω τρόπο δεν θα επιστρέψουμε στην εξάλληψη των ειδών και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα στρέφομαι προ τον Επίτροπο. Έχετε το λόγο λοιπόν κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Για μία ακόμα φορά θέλω να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη για τα σχόλια, τις ερωτήσεις τους που δείχνουν ότι υπάρχει κοινό έδαφος ώστε να προχωρήσουμε την πρόταση αυτή. Εκτιμώ επίσης ότι υπάρχει γενική υποστήριξη από τα αξιότιμα μέλη ε, του σώματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει, όπως κάνατε και όλοι εσείς, την ευαίσθητη φύση του τόνου στα διεθνή φόρουμ και επίσης την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θέλει να συνεισφέρει ε, το τελευταίο μέρος των ποσοστώσεων που έχουμε, το μεγάλο μέρος της ποσότητας που έχουμε, έχουμε και την ευθύνη να έχουμε το μεγαλύτερο μέρος ε, αριθμοφορέων, πράγμα που σημαίνει ότι παίζουμε σημαντικό ρόλο στη διαχείριση αυτού του σημαντικού αποθέματος. Η πρόταση αυτή είναι βασική για την ε, μεταφορά και πάλι ε, των αποφάσεων της ICAT το κοινοτικό δίκαιο. Ο κανονισμός που θα προκύψει θα εξασφαλίσει την νομική βεβαιότητα όσον αφορά τις υποχρεώσεις των φορέων και ως εκ τούτου θα διευκολύνει την εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης της Ένωσης με τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Θα ήθελα να διατρέξω κάποιες από τις παρατηρήσεις που έγιναν. Κυρίως σχεδόν όλοι υπογραμμίζουν το ρόλο της βιοτεχνικής αλίας. Πράγματι, σε μεγάλο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται όπως και το Κοινοβούλιο ε, για τη διατήρηση των ε, παραδοσιακών ε, μέσων αλίας και επίσης μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να υπάρχει παρανόηση στην, στο σχέδιο αλλά βεβαίως ο τόνος δεν είναι δεν είναι το μοναδικό είδος που προσφέρει θέσεις εργασίας και αυτό φαίνεται και από τις ε, ε, προτινόμενες τροπολογίες του κυρίου Μάτο. Θα συμφωνήσουμε να δώσουμε επιπλέον ποσοστώσεις ή να κάνουμε μια ε, μια κατανομή των ποσοστώσεων με άλλο τρόπο. Πιστεύω πως ναι, αυτό μπορεί να γίνει ε, ανακράτος μέλος. Τώρα, έγιναν κάποια συγκεκριμένα σχόλια από ορισμένου ομιλητέ για το αρματράμπα που ανέφερα, που έχει σχέση με τη βιοτεχνική αλία, που πρέπει να προχωρήσουμε τρόπο περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον και πιο βιώσιμο ένας ομιλητής επεσήμανε την σημασία των αποθεμάτων αυτών για τους Ευρωπαίους αλληλείς και πιστεύω ότι πράγματι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Πολλοί από εμά αναφερθήκαμε στις κοινωνικές και οικονομικές πλευρές και θεωρώ ότι η σωστή διαχείριση είναι ο μοναδικός τρόπος να προχωρήσουμε για να προστατεύσουμε τη βιωσιμότητα και την μακρόχρονη βιωσιμότητα των, των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων. Ε, συμφωνώ με την κυρία Ροδούς που είπε ότι οι ποσοστώσει θα πρέπει να είναι διαφανείς κλπ. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει, στο οποίο θα πρέπει να στοχεύουν τα κρέτη μελη και επίσης το θέμα της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Η μικρή κλίμακας βιοτεχνική αλία έχει ρόλο να παίξει σε όλα αυτά. Συμφωνώ με πολλούς από εσά επίσης, οι οποίοι είπατε ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τα πράγματα δεν είναι όσο καλά όσο θα θέλαμε και γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχει περιθώριο ε, αδράνειας. Βεβαίως έχουμε, έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά πολλά ακόμα μένει να γίνουν αναφέρθηκε στον, στον ομοιόμορφο και δίκαιη βάση και την περισσότερη κατανομή προς τους μικρούς αλληλείς. Αναφέρθηκα στο θέμα του σχεδίου διατήρησης για το γάδο. Πιστεύω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε. Τώρα όσον αφορά το EIA ε, που ανέφερε ο Σάντος, είναι κάτι που οι επιστήμονες το λαμβάνουν υπόψη αλλά αν χρειαστεί θα πρέπει να δοθεί και εδώ περισσότερη έμφαση. Όσον αφορά στην αναφορά για, την, για τις κατεξουσιοδότηση πράξη, αυτό είναι βασικό στοιχείο της πρότασης, γιατί θα γίνονται πολλές συχνές τροπολογίες, της ICAT και όλες αυτές πρέπει να ε, γρήγορα να μεταφερθούν στο ευρωπαϊκό δίκαιο και μια άλλη ε, νομοθετική διαδικασία δεν θα μας επιτρέψει να το κάνουμε. Ενώ με τις κατεξουσιοδότηση πράξη θα μπορέσουμε να κινηθούμε ταχαίως σε μη ουσιαστικά σημεία των νομοθετικών πράξεων. Αυτό το ανέφερε ο κύριος Καπούτο νομίζω. Τώρα όσον αφορά την ακρίβεια τα θετικά δεδομένα της ανάκτησης πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Έχει σημειωθεί αυτό και ο κύριος Φερέρα αναφέρθηκε στην σωστή κατανομή. Η Ρενάτε Ρενάτου αναφέρθηκε στα αποθέματα και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Πράγματι, οι ποσοστώσεις θα κατανεμηθούν από τα κράτη-μέλη με τρόπο περισσότερο δίκαιο. Υπάρχει διαφάνεια και αντιπροσωπευτικότητα. Τώρα όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Φάραντς, δυστυχώς σήμερα συζητούμε ε, την, τον τόνο και μόνο αυτό το είδος θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι συμφωνώ ότι μόνο εάν Το λαβράκι μου είπε εδώ. Ότι ε, υπάρχουν 800.000 είπατε ε, που ε, ψαράδες με πετονιά είναι 1,3 εκατομμύρια στη Γαλλία και εφόσον αυτοί εποφελούνται θα πρέπει να αναλάβουν και την ευθύνη τους. Όσον αφορά τις προτάσεις που βάλαμε που, που αφορούν το λαβράκι και δεν συζητήθηκαν, ε, δεν συμφωνώ. Έχουμε ζητήσει από όλα τα κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται να καταλήξουν σε ένα ε, συμφωνημένο σχέδιο. Όσον αφορά το παρότι έχει γίνει κάποια πρόοδος για την αποκατάσταση πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή. Άρα λοιπόν συνολικά θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη για την συμμετοχή τους στη συζήτηση και να ευχαριστήσω τον εισηγητή και το σώμα για την πολύ ε, παραγωγική συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε. Ο κύριο Μάτο, εισηγητή, λοιπόν, έχει το λόγο για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ επίτροπε. Κυρίως ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν και με τον ένα ή άλλο τρόπο βελτίωσαν να βελτιωθεί η ποιότητα. Ευχαριστώ επίσης τους συναδέλφους που στην παρέμβασή τους έδειξαν ότι με τη στάση τους απέναντι στον Επίτροπο δεν έδειξαν ιδιαίτερο σεβασμό, πράγμα το οποίο απορρίπτω κάθετα. Ε, ευχαριστώ όμως όλο, όλους γιατί ακούσαμε τις απόψεις τους. Υπάρχουν δύο θεμελιώδη θέματα. Ένα οι ποσοστώσεις. Κάνουμε λόγο ότι πραγματικά εδώ έγινε μεγάλη προσπάθεια από τους αλλοί και τα αποθέματα τα ανέκαμψαν. Και τώρα για τις, ε, για τα, για τις ποσοστώσεις. Το άλλο σημαντικό ε, θέμα είναι πώς θα γίνει η κατανομή των ποσοστώσεων. Για τα κράτη-μέλη αληθεύει ότι δεν είναι το Κοινοβούλιο, δεν είναι η έκθεση αυτή, αυτό το θέμα που μπορεί να μας κάνει να είμαστε οι πιο αποτελεσματικοί. Όμως είναι ένα πολιτικό μήνυμα, ένα σαφές μήνυμα που πρέπει να αποσταλεί για την καλύτερη κατανομή των ποσοστώσεων, να υποφεληθούν οι μικροί αλληλοί να μην ευνοούνται μόνο οι μεγάλοι. Είναι καλό λοιπόν να υποφεληθούν οι μικροί αλληλείς και η προσπάθειά τους. Γι' αυτό συμμεριζόμαστε αυτή τη θέση και την έχουμε συμπεριλάβει ήδη σε ένα συμβιβασμό, σε μια συμβιβαστική πρόταση, στο ίδιο το κείμενο, με μια τροπολογία που πάει πιο πέρα, αλλά επί της ουσίας αυτό που θέλει απλά είναι να υπάρξει μια πιο δίκαια κατανομή ποσοστώσεων. Και μετά έχουμε και ένα πρόβλημα κύριε Επίτροπε. Πολλές φορές ε, για την κατανόηση των κατεκτέλεση, ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων ε, αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Δεν είναι υπόδειγμα της ταχείας εφαρμογής αυτή η κατάσταση από πλευρά της Επιτροπής και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα ή πρόσχημα αυτή η κατάσταση για να αφαιρεθούν αρμοδιότητες από το Ευρωκοινοβούλιο. Θα μας βρείτε απέναντί σας αν γίνει κάτι τέτοιο. Κάθετα αντίθετους. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, να κάνουμε ό,τι μπορούμε μπορούμε ώστε οι ποσοστώσεις ταχύτατα να μπορούν να εκτελούνται. Σε καμιά περίπτωση όμως ε, δεν θα απεμπολίσουμε τις αρμοδιότητές μας και αυτό πρέπει να κατανοήσετε ως μήνυμα με κάθε σαφήνεια. Είμαι βέβαιος όμως ότι θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περατούτε συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο. Προχωράμε